δείγματα θα κρίνουν όλο το μέλλον αυτού του εγχειρήματος. ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σιγήτρια για την ομιλία σας και για την εργασία που επεταλέσατε. Η διεύρυνση είναι σημαντική για όλους μας. Δεν θα ήμουν πρόεδρος ε, της συνεδρίασής μας αν δεν είχε υπάρξει διεύρυνση. Η διεύρυνση του 2004 συγκεκριμένα. Η διεύρυνση Big Bang. Νομίζω ότι όλοι είμαστε ε, ευχαριστημένοι που θα υποδεχθούμε συντόμως νέα κράτη-μέλη. Η δήλωση του Επιτρόπου με εντυπωσίασε το πώς συνεδίασε την απονομή του βραβείου Νόμπελ με το θέμα που συζητάμε. Νομίζω ότι η ειρήνη, η συμφιλίωση είναι θέματα κλειδιά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγαπητοί συνάδελφοι, κλείνουμε λοιπόν τη συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Το επόμενο θέμα στη ημερήσια διάταξη είναι δήλωση από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής για την κατάσταση στην Κάζα. Θέλω να πιστήσω την προσοχή σας στο ότι μετά από τη συζήτηση δεν θα υπάρξει διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής του Πρόεδρου. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Α, το Συμβούλιο. Με συγχωρείτε, το Συμβούλιο. Ε, yes, ε, ε, excuse me, but in my paper... Με συγχωρείτε. Εδώ έλεγε η Κομισιόν, το Συμβούλιο παρακαλώ έχει το λόγο. Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, είναι η 8η μέρα τη σύγκρουση στη Γάζα, μεταξύ Γάζα και Ισραήλ. Παρακολουθείτε τι εξελίξει, φαντάζομαι. Χθε το βράδυ, ξέρετε τι έγινε. Όλοι είμαστε με την ελπίδα ότι θα υλοποιηθεί η εκεχηρία. Δυστυχώ, οι ελπίδες μας ήταν πρόορες. Γνωρίζω ότι ήταν εν εξελίξει εντατικές διαπραγματεύσεις υπέρ της εκεχηρίας για να ισχύσουν από εχθές τα μεσάνυχτα τοπική ώρα. Η ανακοίνωση της εκεχηρίας αναβλήθηκε. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και σήμερα και είναι ζωτικής σημασίας να καταλήξουν το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε χθε το βράδυ για να συζητήσει τις εξελίξεις και θα συνεχίσει σήμερα αργότερα στη Νέα Υόρκη, εάν αυτό απαιτηθεί. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έλαβα νέα περί τρομοκρατικής επίθεσης ε, κατά λεωφορείου στο Τελαβίβ. Η επαπειραυτή πρέπει να καταδικαστεί με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια. Εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναδιατυπώνει την απερίφραστη καταδίκη κάθε μορφής δηλώσεις και πράξης βίας, ανεξαρτήτως του, από που προέρχεται, ανεξαρτήτως κινήτρου και επαναβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να δώσουμε μάχη κατά της τρομοκρατίας. Η κατάσταση στην περιοχή είναι αβέβαιη, συνεχίζονται επιθέσεις τόσο στο Ισραήλ όσο και στην Γάζα. Εμείς ε, επαναδιατυπώνουμε την έκκλησή μας για αποκλιμάκωση και πάυση των εχθροπραξιών. Οι διπλωματικές προσπάθειες επικεντρωνούν τώρα στην επίτευξη κυχηρίας ως πρώτο μέτρο, πρώτο σταθμό για την εξέβρεση μακροπρόθεσμε βιώσιμη λύση. Προ το σκοπό αυτό είπα ότι εκπρόσωπος και η τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής είναι σε συνεχείς ε, επαφές με τους βασικούς πρωταγωνιστές στην περιοχή αλλά και αλλού. Η κυρία Στον τις τελευταίες ημέρες έχει επαφές με την Αίγυπτο, τις ΗΠΑ, το Ισραήλ, την Παλαιστινιακή Αρχή, τα Ηνωμένα Έθνη και τον Αραβικό Σύνδεσμο κυρία Άστον πρόεδρευση της Υπουργικής στο Κάιρο όπου είχε την ευκαιρία να μιλήσει με βασικούς ε, παράγοντες μεταξύ των οποίων και με τον πρόεδρο Μόρση και τον Αλαραμπή τον γενικό γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου. Είναι σε επαφέ. συνεχής, επαναλαμβάνω, με όλους αυτούς όλες τις τελευταίες ημέρες. Όπως θα έχετε μάθει, Στι 19 Νοεμβρίου, την Δευτέρα, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων κατέληξε στα συμπεράσματα του όσον αφορά την βία στη Γάζα και το Ισραήλ και παραβεβαιώνει τι προσπάθειε να επιτευχθεί εκεχηρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τα εμπλεκόμενα μέρη να πετύχουν εκεχηρία και άμεση αποκλιμάκωση μετά από τα κρούσματα βία ε, τι τελευταίε ημέρε και τις απολύσει αμάχων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ από την λωρίδα της Γάζας τις οποίες ε, είναι υπευθυνή η Χαμάς και άλλες οργανώσεις. Οι επιθέσεις αυτές πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Επίσης τονίζουμε την ανάγκη για όλες τις πλευρές να τηρήσουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Η προστασία των αμάχων ανά πάση στιγμή πρέπει να τηρηθεί αυστηρά. Θυμίζοντας τη στάση μας για τον αποκλεισμό της Γάζας, το κείμενο αυτό αποτελεί ένα συνεντικό κείμενο, ισόρροπο, το οποίο επαναδιτυπώνει την απερίφραστη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κατάσταση. Καραδεικνύει επίσης την ενότητα όλων των κρατών μελών στην παρούσα κρίση. Η κατάσταση στην Γάζα θέτει την Αίγυπτο στο κέντρο των διεθνών προσπαθειών για την επίτευξη λύσης στην κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση την Δευτέρα εξέφρασε την υποστήριξή τη στι προσπάθειες της Αιγύπτου αλλά και άλλων εμπλεκομένων για την επίτευξη ταχαίω εκχειρία. Εκφράζει την ικανοποίησή τη επίση, της καλής υπηρεσίας του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην περιοχή και εκφράζουμε την υποστήριξή μα στην ειρηνευτική του πρωτοβουλία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κάνει ό,τι παίρνει από το χέρι τη για να θερινεί όλε τι πλευρέ να διασφαλίσουν την εφαρμογή και υλοποίηση στην πράξη τη κυρίες και κύριοι βουλευτές, η εκεχηρία είναι προς το συμφέρον και των δύο πλευρών, όχι μόνο υπέρ των αμάχων, οι οποίοι υπέστησαν ήδη σοβαρές απώλειες τις τελευταίες ημέρες. Οι απώλειες ζων αμάχων και στις δύο πλευρές είναι μια τραγική πραγματικότητα, χωρίς να παραγνωρίζουμε και το ψυχολογικό μέρος. Υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα προς τις εξελίξεις στην Γάζα και οι τελευταίες εξελίξεις αποτελούν σαφώς ε, επιδείνωση. Όμως ε, υπάρχει ελπίδα. Τα συνολικά περάσματα στο Κέρελ Σαλόμ παραμένουν ευτυχώς ανοιχτά κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών. Αυτή τη στιγμή τα τρόφιμα ευτυχώ ε, υπάρχουν στην περιοχή. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα διανομής τροφίμων. Δεν έχουν επηρεαστεί επίσης ηλεκτρική ενέργεια, αλλά το νερό και τα φάρμακα ήδη λείπουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίζει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στο ανθρωπιστικό πεδίο και ήδη αφιερώνει μεγάλο μέρος της βοήθειας προς τους Παλαιστινίους, ειδικά στη λωρίδα της Γάζας. Και αυτό δεν είναι μόνο μέσω των Ηνωμένων Εθνών, είναι προσπάθεια περί των προσφύγων, αλλά είναι και απευθείας οικονομική βοήθεια για υπέρ συγκεκριμένων ευάλωτων Παλαιστινιακών οικογενειών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης υποστηρίζει τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες όπως στον τομέα της υγείας και δεσμεύεται να βοηθήσει την Παλαιστινιακή πλευρά για να αναβαθμίσει το πέρασμα στο κ. Μισελόμ, μέσω του οποίου διοχετεύεται κρίσιμη ανθρωπιστική βοήθεια προς την λωρίδα της Γάζας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να επαναργοποιήσει την αποστολή της στην περιοχή μόλις επιτρέψουν οι συνθήκες ασφάλειας για να εισφαλίσει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στο πέρασμα της ράφα όπως ε, άλλωστε συμφωνήσαμε το 2005 για την ελεύθερη διακίνηση. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα του Ισραήλ στην ασφάλεια και παράλληλα η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να απευθύνει εκκλήσεις για την πολιτή. Παύση του όπλων προ την Λωρίδα τη Γάζα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να απευθύνει εκκλήσει για την άμεση και διαρκή άνευ όρων. Άνοιγμα των σημείων διέλευση για εμπορεύματα, φάρμακα και πρόσωπα από και προ την Λωρίδα τη Γάζα. Η θέση τη Γάζας, η κατάσταση στη Γάζα δεν είναι βιώσιμη όσο πολιτικός είναι διαχωρισμένη από την Δυτική Όχθη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναδιατυπώνει την ετοιμότητά τη να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάκαμψη της Λωρίδας της Γάζας σε στενή συνεργασία με την Παλαιστινιακή Αρχή και την Ισραηλινή Κυβέρνηση. Σύμφωνα και με το ψήφισμα 1860 του Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, έκρηξη βία στην Γάζα. συμβαδεύει και σοβαρές πολιτικές αλλαγές στην περιοχή και δείχνει πόσο εύθρευστη είναι η κατάσταση στην περιοχή ακόμη και σήμερα. Θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να επιλύσουμε το Παλαιστινικό. Αυτό θα σταθεροποιήσει την περιοχή και θα αποτελέσει και ανταμοιβή σε αυτούς οι οποίοι τάσσονται υπέρ της περίωσης της βίας. Υποστηρίζουμε τις προσδοκίες του Παλαιστινιακού λαού σε ένα κράτος και, στην, και καταφάσουμε στην ανάγκη του Ισραήλ σε ασφάλεια. Είμαστε υπέρ λοιπόν τη εκεχηρία, η οποία αν εφαρμοστεί με σωστό τρόπο θα βοηθήσει. Όμω δεν θα είναι και επαρκή. Χρειαζόμαστε μια βιώσιμη λύση για την Γάζα και αυτό είναι πιο κατεπίγουσα ανάγκη από ποτέ. Χρειαζόμαστε μια μακροπρόθεσμη λύση η οποία δεν θα επιτρέψει να ξεσπάσει ένας νέος κύκλος βίας. Προς τον σκοπό αυτόν, το σύντομότερο δυνατόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εντείνει τις επαφές της με τους πρωταγωνιστέ στην περιοχή εντός του γνωστού κουαρτέτου αλλά και με τους άλλου παράγοντε, διερευνώντα κάθε δυνατότητα να δημιουργήσει μια νέα δυναμική στην ειρηνευτική διαδικασία. Κυρίε και κύριοι βουλευτέ, μόλι ενημερώθηκα ότι η Αίγυπτος επιβεβαιώνει συμφωνία για εκεχηρία. Θα επιβεβαιώσουμε βεβαίως την πληροφορία, αλλά δεν θέλησα να καθυστερήσω την ανακοίνωση αυτής της πρόσφατης εξέλιξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την αναλυτική πληροφόρηση που μας δώσατε από πλευράς της Προεδρίας, από πλευράς των πολιτικών ομάδων έχουμε διάφορους ομιλητές. Ο κύριος Αλαφράνκα από πλευράς του ΕΛΚ. Δυόμιση λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριοι του Συμβουλίου, κύριε Επίτροπε. Για άλλη μια φορά οι εικόνες ε, της φρίκης ε, μας ε, συγκλονίζουν. Πάνω, και, πάνω από 35 παιδιά πέθαναν τελευταία στη Λοδία της Γάζας. Έξι άτομα εκτελέστηκαν διότι θεωρήθηκαν συνεργάτες του Ισραήλ. Διάφοροι Ισραηλοί πολίτες επίσης πέθαναν λόγω των εκατοντάδων ροκέτων, ρουκετών που ε, εστάλησαν που, στη Λωρίδα της Γάζας από το Ιράν. Είχαμε αυτή την ε, τρομοκρατική απόπειρα στο Τελαβίβ σήμερα και είχαμε επίσης την ε, ε, κινητοποίηση πολλών εφέδρων. Μάθαμε ότι, όπως μας είπε ο Σάλφος Κονμπεντίτ, ότι μετά από τηλεφανήμα των ΗΠΑ και την παρουσία της κυρίας Κλίντον, μετά την κινητοποίηση των Υπουργών της Αραβικής Λίγκας και άλλες εξελίξεις. Είναι προφανές ότι εδώ κύριε Πρόεδρε δεν φτάνουν τα λόγια. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή ότι πέρα από την αδυναμία και τον εκνευρισμό που ε, ε, ε διατυπώνουν τα λόγια του Συμβουλίου των Υπουργών, το σημαντικό είναι να υπάρξει μια κατάπαυση του πυρός που να την εγγυάται ο, Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών και να υποστηρίξουμε έτσι τις πιο μετροπαθείς φωνές. Η εναλλακτική ξέρουμε ποια θα είναι από το 2008 κύριε Πρόεδρε. 1.400 θύματα θρυνήσαμε τότε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι συνθήκες δεν είναι ιδιαίτερα θετικές. Υπάρχει κατακαιρματισμός ε, στις Παλαιστινιακές δυνάμεις, εκλογές στο Ισραήλ τον Ιανουάριο και προφανώς επίσης κλιμάκωση, η πυρηνική κλιμάκωση στο Ιράν. Γι' αυτό, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, αυτό που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασιστικά να υποστηρίξει αυτή η κατάπαυση του πυρός για να αποφύγουμε το χειρότερο. Αλλά να μην ε, γελιόμαστε. Δεν θα υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή. Δεν θα υπάρξει σταθερότητα στην περιοχή την ευρύτερη, ούτε στην ε, ε, στενότερη, εάν δεν αντιμετωπίσουμε τι βαθιές αιτίε και τις αδικίες που προκαλούν αυτή την έκρηξη βία στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Από πλευρά τη Σοσιαλιστική Ομάδα, η κυρία Ντομινίκ Δοκέζα. Δύο λεπτά. Κυρία Πρόεδρε, χαίρομαι για την αναγγελία που κάνετε, κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου, ότι ε, υπάρχει μια κατάπαυση πυρός, αλλά θα πρέπει να κατοχυρωθεί. Αρκετά θύματα θρυνήσαμε μεταξύ του αμάχου πληθυσμού. Αρκετά παιδιά πέθαναν, αρκετό αίμα έχει είναι ανακούφιση αυτό που ακούμε, αλλά νομίζω ότι για να μπορέσει να ισχύσει η κατάπαυση του πυρός πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε και αυτά που λογικά είπε ο πρόεδρος Αμπάς στα Ηνωμένα Έθνη. Γιατί αυτή η τελευταία επιχείρηση του Ισραήλ μοιάζει με την προηγούμενη βεβαίω. Είχαμε την ίδια εγκύτητα με τις εκλογές στο Ισραήλ, την ίδια κλιμάκωση της βίας που από πλευράς Ισραήλ ε, οδηγεί σε εξοδικαστικές δολοφονίες και σε επιθέσεις. Από την άλλη μεριά έχουμε τις ρουκέτες ε, που φεύγουν από την της Γάζας και μάλλον και την απόπειρα σήμερα. Αλλά τώρα κάτι άλλαξε. Δύο. Από τη μία μεριά η Αραβική Άνοιξη που άλλαξε τις διαχωριστικές γραμμές και η Γάζα δεν είναι πια de facto απομονωμένη. Και υπάρχει επίσης και αυτή η επιχείρηση του Ισραήλ, ε, πυλώνας της που είχε ως αποτέλεσμα ε, να σταματήσει να μην θέλει να παρουσιάσει ο, ο, ο Αμπάς τις ε, προτάσεις του στα Ηνωμένα Έθνη. Πρέπει λοιπόν εμείς τώρα ως Ευρώπη να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να υποστηρίξουμε τον πρόεδρο Αμπάς. Η ανησυχία που έχουμε σήμερα για την ασφάλεια του Ισραήλ είναι ουσιώδης. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουμε ευθύνη και για να προσφέρουμε στους Παλαιστινίους μια ε, δυνατότητα κρατικής υπόστασης στα πλαίσια των συνόρων του 67. Είναι ιστορικές και ηθικές αυτές οι υποχρεώσεις μας και βασίζονται στο διεθνές δίκαιο. Στο νότιο, το νότιο Σουδάν μπήκε στα Ηνωμένα Έθνη τρεις μέρες μετά την εξαρτησία του. Ενώ δεν είχαν καθοριστεί ακόμη τα σύνορα και υπήρχε ακόμη πόλεμος με το Σουδάν. Δεν είναι λογικό μετά το 88 από τότε που έχει την ανεξαρτησία της η Παλαιστίνη να εξακολουθεί να είναι στους διαδρόμους του ΟΗΕ. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε όλου του εξτρεμιστέ, όλου αυτού που διαμαρτύρονται για την αδυναμία τη Ευρώπη, που δεν πιστεύουν παρά σε μία λύση μέσω τη βία. Είναι δική μα ευθεία. Δική μα, όχι των ΗΠΑ. Είναι δική μα ευρωπαϊκή ιστορία. Δεν μπορούμε να ζητάμε από του Παλαιστινίου να πληρώνουν τα σπασμένα τη δική μα ιστορία. Με τη Νέα Αίγυπτο, με την οποία ε, διαπραγματευθήκαμε μόλι τώρα φιλόδοξες ε, συμφωνίε, μπορούμε να συνεργαστούμε για να επιλύσουμε την κρίση. Θέλω να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου προ όλα τα θύματα, προ τι οικογένειε όλων των θυμάτων και από τι δύο μεριέ, αλλά δεν θα έπρεπε να πληρώσουμε τη ζωή του, τι ε, ευθύνε μα και την ιστορία μα. Ο πλευρά τη ε, Άλντε, η κυρία Νέιτς Έιτενμπρουκ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Πριν από πάνω από δέκα χρόνια από πλευρά ε, του Νάβιλ του που ήταν ο υπεύθυνο για τις διαπραγματεύσεις της Βρυξέλλες εξ ονόματος των Παλαιστινίων είπε εκφράζουμε τη θλίψη μας για τα θύματα, το αίμα των παιδιών μας. Από τότε δεν σταμάτησε ποτέ η βία δυστυχώς και τα πιο πρόσφατα γεγονότα είναι ιδιαίτερα αιματηρά ουσιαστικά βλέπουμε ότι δεν είναι το πιο σημαντικό να ξέρει κανείς ποιος ξεκίνησε τη βιοπραγία. Όσο πιο πίσω πάει κανείς ε, αλλάζει ο πρωταγωνιστικός ρόλος των υπεύθυνων, των ενόχων και έχουμε αυτό τον φαύλο κύκλο δράσης-αντίδρασης, πράξης και αντεκδίκησης. Ελπίζω βαθιά στην καρδιά μου ότι θα υπάρξει και χειρία τελικά και ότι οι προσπάθειες της Αιγύπτου και όλων των άλλων εμπλεκόμενων ως διαμεσολαβητών θα ευδοκιμήσουν και θα μπορέσουν να οδηγήσουν στο να υπάρξει μια σταθερή εκεχηρία πλέον, διαρκέστερη εκεχηρία. Σε σχέση με τους προλαλήσαντες πρέπει και εγώ να πω ότι πρέπει να προσπαθήσουμε τα αίτια της βίας να τα αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν μπορεί να ζήσει μέσα σε ένα καθεστώς ειρήνης, σε ειρήνη το Ισραήλ και να υπάρχει δίπλα στο Ισραήλ και ένα Παλαιστινιακό κράτος που θα ζει και αυτό σε ειρήνη. Ελπίζω ότι οι μεταβολές που επισυνέβησαν σε όλη αυτή την περιοχή του κόσμου και τα πρόσφατα γεγονότα θα μπορέσουν να οδηγήσουν να αναγνωρίσουν όλοι ότι το status quo δεν μπορεί να συνεχιστεί πλέον διότι δεν υπάρχει αηφορία σε αυτό το καθεστώς, το status quo. Πρέπει με κάθε προσπάθεια να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, να υπάρξει μια μελλοντική προοπτική συμβίωση των Ισραηλινών και των Παλαιστινίων. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Και στη συνέχεια, εξ ονόματος των Πρασίνων, ο κύριος Κον Μπεντιτ, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, είναι η ώρα να πούμε μερικές απλές αλήθειες. Η απλή αλήθεια είναι ότι δεν είναι δυνατόν βομβαρδίζοντα με ρουκέτε στο Ισραήλ ή με τρομοκρατικέ απόπειρε στο Τελαβίβ, θα κατα... δεν πρόκειται να καταλήξουμε έτσι σε παλαιστινιακό κράτο. Δεν είναι δυνατόν συνεχίζοντα του επικισμού. Δεν είναι δυνατόν συνεχίζοντα να μην δίνουμε προοπτικέ στου Παλαιστινίου, θα καταλήξουμε στην ασφάλεια του κράτου του Ισραήλ. Νομίζω ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να αναλάβει τι ευθύνε του. Οι ευθύνε για το Κοινοβούλιο μα είναι να καταδείξει τη στρατηγική που θα μπορούσε να οδηγήσει στην ειρήνη η στρατηγική είναι σαφής. Πρέπει ένα ναι χωρίς καμία επιφύλαξη και απόχρωση ε, στην ε, ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ. Πρέπει ε, επίσης ανεπιφύλακτα να πούμε ναι σε ένα Παλαιστινιακό κράτος. Ένα Παλαιστινιακό κράτος που να μην το περιορίζουν οι επικισμοί. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τη στρατηγική μη βίας του Προέδρου Αμπάς. Εάν δεν υποστηρίξουμε αυτή τη στρατηγική στην πράξη υποστηρίζουμε αυτούς που δεν θέλουν την ειρήνη. Και γι' αυτό είναι πολύ καλό που το ψήφισμα του Κοινοβουλίου που θα ψηφίσουμε αύριο αναφέρει συγκεκριμένα, εκπεφρασμένα, ότι υποστηρίζουμε τη στρατηγική του Προέδρου Αμπάς να απευθυνθεί στον ΟΗΕ και να ζητήσει την αναγνώριση καθεστώτος παρατηρητού για το Παλαιστινιακό κράτος. Αν δεν το κάνουμε αυτό, αν δεν ζητήσουμε να αρθεί ο αποκλεισμός της Γάζα με διεθνή έλεγχο, τότε δεν θα καταλήξουμε σε ειρήνη στην περιοχή. Δεν μπορούμε να αποκλείουμε 1,5 εκατομμύριο Παλαιστινίους και να θεωρήσουμε ότι θα μείνουν λογικοί και φρόνιμοι. Είναι τρομερό αυτό που κάνει το Ισλαμικό Τζιχάντ. Είναι τρομερό να εκτοξεύονται πύραυλοι κατά του Ισραήλ. Πρέπει να σταματήσει, αλλά δεν θα σταματήσει παρά μόνο εάν αυτοί οι άνθρωποι στη Γάζα έχουν μία προοπτική για τη ζωή του. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να το κατανοήσει κανεί αυτό και γι' αυτό τονίζουμε ναι στην ειρήνη του Ισραήλ, ναι, ναι στην ασφάλεια του Ισραήλ, ναι στην ταυτότητα του Ισραήλ, ναι στην Παλαιστίνη, να σταματήσει ο αποκλεισμό και να υποστηρίξουμε τον πρόεδρο Αμπά στον ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενος ομιλητής. Μισό λεπτό. Παρακαλώ, είστε έτοιμοι να, να μιλήσετε. Α, ε, υπάρχει μία μπλε κάρτα. Ε, είστε διατεθειμένος να δεχτείτε. Βεβαίως, παρακαλώ. Παρακαλώ. Θέτω το ερώτημα. Κύριε Γκόλπεντιτ, νομίζετε ότι η προσπάθεια να ανοίξει για οικονομική και ανθρωπιστική βοήθεια η λωρίδα της Γάζας είναι να το να γίνει αν δεν σταματήσουμε και την εισαγωγή κυρίως από το Ιράν πυράβλων και άλλου στρατιωτικού υλικού. Ευχαριστώ πολύ. Κονπεντήτ. Αγαπητέ συνάδελφοι, θα σας έλεγα νομίζετε ότι ο αποκλεισμός της Γάζας Εμπόδισε την είσοδο πυράβλων. Όχι. Την απόδειξη την έχετε. Έχουν εκτοξεύσει, ενώ υπάρχει αποκλεισμό πάνω από χίλιε. Θα ήταν ίσω πιο ευφυέ και από τη δική σα την πλευρά να επιχειρήσετε να καταλάβετε ότι σήμερα ένα αποκλεισμό ή μάλλον η άρση του αποκλεισμού με διεθνή έλεγχο, ούτω ώστε να ε, ε, εισαχθούν οικοδομικά υλικά να εισαχθούν ε, τα υλικά της ανθρωπιστικής βοήθειας, αυτό θα βοηθούσε και θα ελεγχθούν τα άλλα. Εάν δεν υπάρχει επαρκής διεθνής έλεγχος, θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα υπόγεια περάσματα για να εισάγονται οι, ροκε, ρουκέτες. Και ο πληθυσμός της Γάζας θα είναι όλο και πιο πολύ απεγνωσμένος. Ευχαριστώ. Επόμενος μιλητής, εκ μέρους της ομάδας CCR, είναι ο κ. Στανόκ. Πρόεδρε, άλλος μίλησε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Οι επιθέσεις, οι τελευταίες είναι μια ανθρώπινη τραγωδία. Προκλήθηκαν από τις εκτοξεύσεις ρουκετών, καταρχήν, κατά του Ισραήλ, στοχεύοντας αδιακρίτως αμάχους σκοτώνοντας πολλούς από αυτούς και καταστρέφοντας υποδομές. Κάθε κράτος, βάσει του άρθρου 51 των Εθνών έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Καλώς λοιπόν το Ισραήλ ερμητοποιήσει την κατάσταση και καταστρέφει εκτοξευτήρες και οπλοστάσια. Οι εκτοξευτήρες βρίσκονται σε περιοχές κατοικίας, κάτι το οποίο αποτελεί ένα άλλο έγκλημα πολέμου. Η ομάδα βεβαίως υποστηρίζει τα δύο κράτη βάσει ενός βιώσιμου κράτους της Παλαιστίνης, το οποίο θα ζει ειρηνικά με το Ισραήλ. Όμως τέτοια προοπτική δεν υπάρχει όσο την Γάζα τη φεδεύουν τορμοκράτες οι οποίοι θέλουν να καταστρέψουν το κράτος του Ισραήλ. Και φυσικά θέλουμε να δούμε διαπραγματεύσει, να, να ξεκινήσουν διαπραγματεύσει υπό τον μετροπαθή Αμπά. Όμω δεν με πείθουν οι σχετικέ ε, επικλήσει. Ούτε πείθομαι επικλήσεις για την άρση του αποκλεισμού, διότι οι πολιτικές ε, εγγυήσει δεν μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα συνεχιστεί το λαθρεμπόριο όπλων, κυρίως μέσω του Ιράν για θαλάσσεις. Εκφράζω τη συμπαραστασή μου στα σημερινά θύματα, 10 τραυματίες στο Τελαβίβ, κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι θα επιτρέψει στις Αιγυπτιακέ επικλήσει να πετύχουν. Χαίρομαι όμω για τα νέα που μόλι ε, ανακοίνωσε η Υπουργό Εξωτερικών τη Κύπρου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τάνοκ. Έχουμε μια μπλε κάρτα. Ε, είστε έτοιμο να απαντήσετε. Πάντα. Κύριε Πρόεδρε, κύριο Μέρφυ, παρακαλώ. Ο φίλο μου κύριο Μέρφυ, από την αντίθετη πλευρά. Κύριε Τάνοκ, πιστεύετε πραγματικά ότι η επίθεση κατά του πληθυσμού της Γάζας σχετίζεται με την προστασία του Ισραηλινού λαού. Δεν βλέπετε την σχέση μεταξύ αυτών των επιθέσεων και των προσεχών εκλογών τον Ιανουάριο στο Ισραήλ. Δεν βλέπετε ότι η τελευταία έκρηξη μεταξύ άλλων είχε ω θύμα ένα 12χρονο παιδί που έπαιζε απλώ ποδόσφαιρο στη Γάζα. Και πώ εξηγείται τα χειρουργικά πλήγματα με τα οποία βρήκαν το θάνατο 150 Παλαιστίνη, οι περισσότεροι ε, άμαχοι. Πόσο, χειρουργικά είναι λοιπόν αυτά τα πλήγματα. Απάντηση. Η διαφορά είναι ότι το Ισραήλ δεν ε, πλήττει αδιακρίτως αμάχους όπως ε, η Χαμάς όταν εξαπολύουν ρουκέτες κατά του Τελαβίβ και της Ιερουσαλήμ. Καταστρέφουν στρατιωτικούς στόχους οι Ισραηλοί. Και φυσικά κάθε παιδί που χάνεται, κάθε γυναίκα είναι μια τραγική απώλεια. Όμω ο στόχο δεν είναι ο θάνατο των αμάχων, είναι να καταστραφούν οι εκτοξευτήρε των ρουκετών και οι υπεύθυνοι. Σε καμία περίπτωση λοιπόν ο στόχο δεν είναι η καταστροφή τη Λωρίδα τη Γάζα. Ο κ. Τάνοκ φαντάζομαι θα απαντήσει και την επόμενη μπλε κάρτα. Μισό λεπτό παρακαλώ. Πάντα θαυμάζω το πόσο καλά γνωρίζετε και κατανοείτε τα θέματα για τα οποία κάνετε λόγο. Τώρα ωστόσο όμως αναφέρατε κάποια γεγονότα σαν να ήταν κάποιες ασκήσεις σκοπευτών στη Μέση Ανατολή. Θα ανέμενα και σας ζητώ κιόλας να πείτε δεν πιστεύετε ότι αυτά τα πρόσφατα γεγονότα θα έπρεπε να μας υπενθυμίζουν ότι θα έπρεπε να εξευρεθεί μια δίκαια πολιτική λύση στα προβλήματα της Μέσης Ανατολής και να ξεκινήσουν επιτέλους σοβαρές διαπραγματεύσεις με βάση την αρχή δύο κρατών που θα συμβιώνουν ειρηνικά μεταξύ τους. Κύριε Τάνοκ, το κατέστησα σαφέστατο στη δική μου παρέμβαση. Φυσικά είμαι υπέρ της λύσης των δύο ξεχωριστών κρατών για το Ισραήλ και την, τους Παλαιστίνιους με ένα Παλαιστινιακό κράτος που θα ζουν ειρηνικά και θα συμβιώνουν το ένα κράτος δίπλα στο άλλο. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι η πάυση των τρομοκρατικών πράξεων κατά του Ισραήλ από τους Παλαιστίνιους και να μπορέσουν οι Ισραηλινοί να θεωρήσουν ότι μπορούν να προσέσουν σε διαπραγματεύσεις υπό την αιγίδα της τετραμερούς. Αυτή τη στιγμή όταν πύραυλοι εκρήγνυνται στην επικράτειά τους δεν έχουν καμιά εμπιστοσύνη στην ιδέα αυτή της συνύπαρξης των δύο ξεχωριστών κρατών. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ και εξ ονόματος στη συνέχεια της ε, ομάδας υπέρ της, ε, των ελευθεριών της δημοκρατίας ο κύριος Μπέντερ. Σας ευχαριστώ. Μία παρατήρηση θα ήθελα να κάνω. Η συζήτηση για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας ε, θα πρέπει να μας κάνει να δούμε την κατάσταση στο Ισραήλ και τη Λωρίδα της Γάζας από κοινού, διότι η της Χαμάς που πέφτουν στο Ισραήλ και των ε, τζιχαντικών ομάδων οδηγούν σε αυτήν την έκρηξη βίας ε, που σημειώνεται σε σχέση με το πρόβλημα της Λωρίδας της Γάζας. Υπερασπίζονται τη ζωή τους ε, και τα αγαθά τους, την περιουσία τους στο Ισραήλ και αυτό βαίνει καλώς και είναι δίκαιο. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι καμιά φορά δυσανάλογα ακολουθούνται κάποιες δράσεις και γι' αυτό υπάρχει κλιμάκωση της βίας. Τρία στοιχεία εμπεριέχονται εδώ σε, αυτό το, σε αυτή την πρόταση ψηφίσματος. Ελευθερία για τους Εβραίους, τους Παλαιστίνιους σε σχέση και με την Ιερουσαλήμ. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να τοποθετηθούν επ' αυτού σε σχέση με την έκρηξη βίας στη Λωρίδα της Γάζας. Θα πρέπει με κάθε τρόπο, με ό,τι περνάει από το χέρι μας να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να αποσοβηθεί ο κίνδυνος που ε, υπάρχει κατά του Ισραήλ και σε σχέση με την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Κατάρ θα έπρεπε να υποστηρίξουν αυτή την κοινή προσπάθεια. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ για την Ευρωπαϊκή Αριστερά. Ο κύριος Λεχιαρίκ, τρία λεπτά παρακαλώ. Είναι τόσο λυπηρή αυτή η κατάσταση, τόσο επώδυνη η κατάσταση. Πρέπει η πολιτική να αντιμετωπίσει, να αντικαταστήσει τη βία. Το κοινοβούλιο μας πρέπει να ψηφίσει ένα σαφές ψήφισμα, ένα ισχυρό ψήφισμα για να υποστηρίξουμε την κατάπαυση του πυρός, εάν υπάρχει, για μια διαρκή ειρήνη, για την επίλυση μέσω δύο κρατών. Αλλά πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο τις δύο πλευρές σε αυτήν την ε, υπόθεση υπάρχει ένας επικιστής και ένας ε, επικιζόμενος. Στο λόγο της Γκάζας επιβάλλεται από κάποιον άλλον κάποιος αποκλεισμό. Καταδεικνύοντας ε, τον Χαμάς ως τον κύριο συνομιλητή μας αποδυναμώσαμε τον, την οργάνωση για την απελευθέρωση Παλαιστίνης που εδώ και 20 χρόνια έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία διαλόγου η διεθνή κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποδυνάμωσαν και ταπείνωσαν την Παλαιστινική Αρχή και επίσης αποδέχονται πλήρη ασυδοσία των Ισραηλινών υπευθύνων. Ποτέ δεν πήραμε καμία πολιτική απόφαση για να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο. Αυτό τροφοδοτεί τις ακραίες ομάδες που αυτή την απαράδεκτη πολιτική του επικισμού, του πολέμου και του αποκλεισμού την αξιοποιούν. Όπως και πριν από τέσσερα χρόνια, οι θύνοντες ε, του Ισραήλ ξεκινάνε ένα πόλεμο, κάνουν πολιτική φόβου και αίματος με ε, στόχο την προκλογική εκστρατεία. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η στρατιωτική, η, στρατι, επιχείρηση θέλει να παρεμποδίσει το καθεστώς παρατηρητή του Παλαιστινιακού κράτους. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να γίνει σεβαστό το διεθνές δίκαιο και μπορούμε να το κάνουμε αξιοποιώντας το άρθρο 2 της Συμφωνίας Σύνδεση μπορούμε να το κάνουμε υποστηρίζοντα σαφώ τι προσπάθειε του Μαχμούτα Αμπάς για να αναγνωριστεί για την Παλαιστίνη η ιδιότητα συνδεδεμένου μέλου. Δεν υπάρχει πιο συγκινητική κραυγή από εκείνη τη κυρία Μισελ Βασέρ, που είναι μια Ισραηλινή που ζει τρία χιλιόμετρα από τα σύνορα τη Γάζα, που την απέστειλε στην, ε, στον Πρωθυπουργό και που δημοσιεύτηκε στη Χαρέτ. Και κάνω παραπομπή. Εάν ε, ενδιαφέρεστε για μα, σταματήστε να μας ε, υπερασπίζεστε με πυράβλους. Αντί για την επιχείρηση πυλώνας της άμυνας, ξεκινήστε την επιχείρηση ελπίδα για το μέλλον. Συμφωνώ απόλυτα με τα λόγια αυτά, γιατί δεν θα μπορούσα να πω τίποτα καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κύριος Μπέλτερ σήκωσε μια μπλε κάρτα. Θα θέλατε να την δεχτείτε την ερώτηση και να απαντήσετε. Έχετε τον λόγο κύριε Μπέλντερ, παρακαλώ. Ο κύριος Μπέλντερ. Ναι, αγαπητέ συνάδελφε Γερίκ, ακριβώς όπως και σε σχέση με τον σύντροφο, από, σύντροφό σας από την Ιρλανδία, πιστεύω ότι μια διασύνδεση δημιουργείται μεταξύ της κλιμάκωσης της βίας και των εκλογών στο Ισραήλ. Μια ερώτηση θα είχα. Πώς μπορείτε αυτό να το τεκμηριώσετε και να το αποδείξετε με γεγονότα και ε, πραγματικά τεκμήρια, διότι είναι ένας ισχυρισμός αυτός, αβάσιμος, που δεν ε, τεκμηριώνεται από κανένα γεγονός. Διότι όποιος γνωρίζει την κατάσταση στη Μέση Ανατολή γνωρίζει πώς υπήρξε η κλιμάκωση της βίας. Η Χαμάς ήταν εκείνη που συνεργάζεται με την Αλκάιδα σε σχέση με την Λωρίδα της Γάζας. Θα ήθελα να ακούσω ποια είναι τα τεκμήρια που έχετε, διότι αυτό είναι ένας αβάσιμος ισχυρισμός. Το που λέτε είναι απόλυτα λάθος. Πρώτον, εδώ και τέσσερα χρόνια η ΑΜΑΣ παίζει ρόλο μετριοπαθή και προσπαθεί να εφαρμόσει την εκεχηρία. Υπάρχουν ε, άλλες ομάδες όπως το Ισλαμικό Τζιχάντ, ακραίες, που προκάλεσαν ή έχουν προκαλέσει ορισμένε φορές την εκτόξευση ε, πυράβλων και ρουκετών. Το γεγονός ότι δολοφονήθηκε ο επικεφαλής στρατηγικής ομάδας του Χαμάς που είχε διαπραγματευθεί ανταλλαγή εχμαλώτων και διαπραγματευόταν ε, εκεχηρία ήταν η πράξη που δημιούργησε την κλιμάκωση. Επαναλαμβάνω ότι αυτό όπως και πριν από τέσσερα χρόνια γίνεται παραμονές των, των Ισραηλινών εκλογών. Παρακαλώ, έχει το ε, λόγο για ένα λεπτό. Καλωσορίζω τις ε, πληροφορίες για μια ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Πιστεύω ότι όλοι ενωμένοι πρέπει να χαιρετήσουμε αυτή την εξέλιξη που μόλις μας παρουσιάστηκε. Ελπίζω αυτή η κατάπαυση του πυρός να φέρει κάποια σταθερότητα σε μια πολύ εντεταμένη και ε, βίαιη κατάσταση. Πρέπει επίσης όλοι μαζί να καταδικάσουμε την τρομοκρατική απόπειρα κατά του λεωφορείου στο Τελαβίβ. Πρέπει να υπερασπιστούμε το δικαίωμα του Ισραήλ να προστατεύει όλους τους πολίτες από επιθέσεις με πυράβλους. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε το ρόλο του σώματός μας και των θεσμικών μας οργάνων. Δεν νομίζω ότι έχουμε κατά νου τον κύριο στόχο. Έχουμε επιτρέψει πολλούς μήνες να γίνονται αυτές οι επιθέσεις με ρουκέτες επανειλημμένα κατά του Νότιου Ισραήλ από τη Γάζα και μόνο όταν γίνει τόσο τεταμένη η κατάσταση, τόσο βίαιη, ασχολούμεθα με αυτό. Πρέπει να παίξουμε το ρόλο, το ρόλο έντιμου διαμεσολαβητή σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να μην επιδιώκουμε καθεστώς κράτους στα Ηνωμένα Έθνη, αλλά να επιδιώξουμε τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και μία μακροπρόθεσμη λύση. Μπλε κάρτα. Ε, θέλετε να απαντήσετε. Ναι. Παρακαλώ. Όσον αφορά την ασφάλεια του Ισραήλ και την άμυνα των πολιτών του. Για να γίνει αυτό, Πιστεύετε ότι είναι ρεαλιστική ελπίδα όταν αναβάλουμε την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτου, όταν γνωρίζουμε τα δημογραφικά δεδομένα στην περιοχή και όταν τα στοιχεία αυτά είναι κατά της ασφάλειας του Ισραήλ, εάν τα πράγματα φυσικά συνεχίσουν να είναι όπω είναι σήμερα. Ευχαριστώ τη συνάδελφο για την ερώτηση. Γνωρίζω την ειρηνευτική διαδικασία στην περιοχή μου και να σας πω ειλικρινώς ότι για να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμη σταθερή ειρήνη, χρειάζεται εμπιστοσύνη. Δεν νομίζω ότι οικοδομούμε την εμπιστοσύνη επιδιώκοντας άλλους σκοπούς, άσχετους σκοπούς, ενώ το ζητούμενο είναι, επαναλαμβάνω, η αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ας δούμε τι χρειάζεται το Ισραήλ για να ξανακαθίσει το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όπω φυσικά πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το οποίο ακριβώς ε, ζητούν οι Παλαιστίνοι. Το θέμα και πάλι είναι η εμπιστοσύνη και ο ρόλος του έντιμου διαμεσολαβητή για να διασφαλίσουμε ότι εφαρμόζουμε ίδια μέτρα και ίδια, ίδια σταθμά προς τις δύο πλευρές. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και τώρα για να καταλήξουμε εγκατακλείδει η Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, μπορώ να επιβεβαιώσω ότι όντως συνεφωνήθη η κατάπαυση του πυρός όπως ε, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μοχάμετ Άμαρ και η κυρία Χίλερη Κλίντον, Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου πριν από λίγα λεπτά. Η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ στις 7 ε, η ώρα, ώρα Greenwich. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, με τη συζήτηση περί των εξελίξεων στην Γάζα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέδειξε για άλλη μια φορά την βαθύρατη και γνήσια ανησυχία του για τους αμάχους στην περιοχή, καθώς και την διαρκή του υποστήριξη στην επίτευξη βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. 130 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο στην Γάζα και 5 στο Ισραήλ μέχρι χθε το βράδυ. Πολλοί από αυτού είναι αθώα θύματα, γυναίκες και παιδιά. Είχαμε και επιπλέον θύματα σήμερα στη Γάζα. Οφείλουμε σε αυτούς τους ε, αθώους ανθρώπους να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να δοθεί η μόλις επιτευχθήσα κατάπαυση του πυρός. Και βεβαίω η ειρήνη ε, και το τέλος της, του αποκλεισμού της λωρίδας της Γάζας. Απευθύνω και πάλι έκκληση στο Ισραήλ να φροντίσει για την προστασία των αμάχων. Επίσης, αποδοκιμάζω τις συνοπτικές εκτελέσεις 7 Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας τις τελευταίες μέρες από ομάδες ενόπλων της περιοχής. Αυτό αποτελεί την πλέον κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Η συμφιλίωση και μεταξύ των Παλαιστινίων παραμένει ένα ουσιώδες στοιχείο, μια ουσιαστική ανάγκη για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης. Και πρέπει να μην ξεχνούμε ότι η κατάσταση στην Γάζα είχε επίσης ως αποτέλεσμα ένταση και στην όχθη με δύο νεκρούς κατόπιν διαμαρτυριών στις 18 και 19 Νοεμβρίου. Η ενότητα των Παλαιστινίων είναι άλλο ένα σημαντικό στοιχείο για να οδηγηθούμε προς ένα βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος και για βιώσιμη ειρήνη με το Ισραήλ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαρκώς απευθύνει σχετικές εκκλήσεις. Ο πρόεδρος Αμπάς προσπάθησε προς την κατεύθυνση αυτή και νομίζω το ίδιο και η Αιγύπτιοι από την υπογραφή της συμφωνίας τον Μάιο του 2011 για τη διαπραγμάτευση της σύμβαξης δύο κρατών την οποία υποστηρίζουμε. Αυτή ακριβώς αποτελεί και την μόνη βιώσιμη λύση για τον Ισραηλινό λαό και τους Παλαιστινίους. Η κλιμάκωση της βίας, ως αυτή που παρατηρήσαμε τις τελευταίες ε, ημέρες, αποτελεί μια τραγική παρέκβαση από την πορεία που πρέπει κανονικά να ακολουθήσουμε. Ευχαριστώ. σε ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κάποτε, μια φορά και έναν καιρό, στη σοβιετική σφαίρα επιρροής, όπως την